Συζητάμε στα θέματα των ε, ε, ημερησίων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουμε μία ώρα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας και καταρχήν έχουμε το θέμα της Νοτιοαφρικής ε, σφαγή απεργών ανθρακορίχων και η συζήτηση ξεκινά με την κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να δούμε με προσοχή αυτό το θέμα, διότι όταν υπάρχουν 58 τραυματισμένοι και 38 νεκροί και πολλοί από αυτούς είναι ανήλικοι, εγώ αυτό το ονομάζω σφαγή. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενοχλεί είναι ότι πρόκειται για μια φίλη χώρα. Χώρα που έχει αγωνιστεί κατά το Απαρτχάιτ και η Νότιος Αφρική είναι κάπως ε, τροποντινά ένα πρότυπο. Αλλά ακόμα και με τέτοιε χώρε που μπορεί να αποτελούν πρότυπο, που είναι φίλε, θα πρέπει να μπορούμε να πούμε την αλήθεια. Νομίζω ότι ο πρόεδρο τη χώρα το έχει καταλάβει. Έχει ξεκινήσει μια έρευνα, η οποία μπορεί να ξεκινήσει άσχημα, <coughs> διότι οι μεταλλορίχοι, οι οποίοι απεργούσαν κατά των απαράδεκτων συνδικών εργασία, ε, ήταν θύματα ή απειλούνταν με δολοφονία. Εδώ λοιπόν πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει κάποια δέσμευση στις σχέσεις μας με τις χώρες της Αφρικής. Θα πρέπει να ασχολούμαστε πολύ σοβαρά και με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων που έχουν μετατοπιστεί εκεί. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο αισθανόμαστε συνυπεύθυνοι για όσα συνέβησαν στην Αφρική. Ευχαριστώ. Επόμενο μιλήτρια η κυρία Κιλ Νίλσεν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, ε, αισθανόμαστε ότι πρέπει να αρθούμε εναντίον ε, αυτής της αιματηρής κατάστασης η οποία θυμίζει μαύρες σελίδες της ιστορίας της Νοτιοαφρικής. Πρέπει να υπάρχει ε, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό και χαίρομαι ότι υπάρχει μία εξεταστική επιτροπή η οποία θα εξετάσει τα γεγονότα της 16ης Αυγούστου αλλά θα πρέπει συνήθως ε, να ε, καταδικάσουμε την προσφυγή η οποία θυμίζει την νομοθεσία η οποία θυμίζει την εποχή της Υπάρχει μεγάλη φτώχεια σε ένα μέρος του πληθυσμού και εξού και οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να αλλάξει η κατάσταση και αντιθέτως διαπιστώνουν ότι υπάρχει μία νέα οικονομική apartheid. Ε, το θέμα αυτό παραμένει πολύ σημαντικό για την ε, ε, Νότιο Αφρική εξού και η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει μία μία διαφορετική κίνηση σε αυτή την περιοχή και να απαγορεύσει την εξαγωγή των ορυκτών προϊόντων τα οποία εξορίζονται χωρίς σεβασμό των, ε, του περιβάλλοντος. Επιπλέον πλέον της δημοκρατίας χρειάζεται και περισσότερο κοινωνική δικαιοσύνη στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τάνοκ για ένα λεπτό. Έχουν περάσει δύο δεκαετίε από τον τερματισμό του Απαρτχάρτ και τι πρώτε δημοκρατικέ εκλογέ στην Νότια Αφρική και έχει κάνει τεράστια άλματα η χώρα αυτή. Έχει μεγάλη οικονομική δύναμη. Γι' αυτό έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί σωστά και τα κοιτάσματα χρυσό που διαθέτει. Θα πρέπει όμω να σκεφτούμε ότι η αφρικανική πολιτική, η πολιτική μάλλον τη Νότια Αφρική, με τις γειτόνες χώρες μπορεί να είναι φιλική, όμως εσωτερικά φαίνεται να υπάρχουν εδώ προβλήματα με την εκπαίδευση της αστυνομικής ε, δύναμη λόγου χάρη, που δεν είναι επαρκή ε, και υπάρχουν πολλές παραβιάσεις δικαιωμάτων. Εδώ λοιπόν, εκ μέρους τη ομάδα μου, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας προ τους, προς τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματισμένων ε, απεργών. Όμως, ο πρώην ο πρώην ε, αρχηγός της νεολαίας ε, στη Νότια Αφρική έχει καταληφθεί την κατάσταση αυτή. Για πολιτικούς σκοπούς αυτό απειλεί την σταθερότητα και την ειρήνη στην Νότια Αφρική. Την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστούμε. Δυστυχώς έκανα ένα λάθος. Η κυρία Βερζιά είναι επόμενη για ένα μισή λεπτό. Δεν θα σας ε, ο Πρόεδρε, γιατί η Γκουε θα πρέπει να είναι τρίτη, αλλά δεν πειράζει. Το τέρμα του Απαρτχάιτ και η ανάληψη τη εξουσία από τον κύριο Μαντέλα το 1994 ήταν πραγματικά ένα μεγάλο βήμα για ολόκληρο τον κόσμο. Όμω 15 χρόνια αργότερα, για εκατομμύρια νοτιοφρικανών, η ελπίδα χειραφέτηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Μετά από πολλά χρόνια ε, προσπαθειών η Νότια Αφρική έχει συμμετάσχει στη δικασία παγκοσμιοποίηση και στην ε, διεθνή οικονομική εξέλιξη, αλλά με τι τίμημα. Βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ε, Νοτιοαφρικανών που μοιράζονται τα πλούτη τη χώρα αυτή, ενώ το 58% του πλούτου συγκεντρώνεται στα χέρια των λίγων, που είναι λευκοί και ελάχιστοι μαύροι. Ναι, υπάρχει οικονομικό απαρτιχάιτ πλέον στη χώρα αυτή. Και όλα αυτά έχουν ένα τίμημα. Ε, η απεργία του φετινού καλοκαιριού στα ορυχεία της Μαρικάνα αφορούσε μεταλλορύχους, λευκούς και μαύρους και έχει δείξει ότι είναι κοινωνική διάσταση η αποτυχία της χώρας αυτής. Δεκάδες νεκροί, ε, χάρη στην ε, τόσο εσφαλμένη παρέμβαση της αστυνομικής ε, δύναμης και τελικά και με τη δικαστική παρέμβαση τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν. Πρέπει να αντιδράσουμε λοιπόν. Θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν πρόκειται για ένα απομονωμένο γεγονό. Μόνο το 2010 η βία τη αστυνομία οδήγησε σε 1.500 θανάτου περίπου. Η, το ισόρροπο ψήφισμα που πρέπει να εγκρίνουμε θα πρέπει να, να συμβάλλει στην αλλαγή αυτή τη κατάσταση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πόσελ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, είμαι πολύ ευγνώμων που ε, όλοι ζητούν ε, να υπάρξει ε, πλήρης σαφήνεια σχετικά και διαφάνεια σε αυτή την αιματοχυσία και θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί του κειμένου και όχι μόνο στην επικεφαλίδα γι' αυτό και είμαι σαφής και ευχαριστημένος που έχετε τοποθετηθεί έτσι. Θέλουμε να στηρίξουμε τη Νότιο Αφρική που για μας είναι ένα σημαντικός εταίρος και που έχει υποφέρει πάρα πολύ από το καθεστώς της Απαρτάιτ και οι Ευρωπαίοι είναι συνυπεύθυνοι. Τώρα όμως πρέπει να μην αποδυναμωθεί η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα και δυστυχώς βλέπουμε ότι εδώ δεν πρόκειται για μία μεμονωμένη περίπτωση ή για ένα τύχημα αλλά ενδεχομένως για μία συστηματική εξέλιξη ε, για τον εκδημοκρατισμό και ε, αυτό, αυτή είναι η σημασία αυτού του ψηφίσματος. Εδώ, κυρία Όγλαντ, οι πυροβολισμοί και οι τραυματισμοί απεργών από τις 16 Αυγούστου είναι ένα τραγικό γεγονός ένα τραγικό σφάλμα των νοτιοαφρικανικών αρχών. Είναι ένα τεράστιο σφάλμα κρίσης και οδήγησε σε τεράστιε διαδηλώσει και διαμαρτυρίες. Η απεργή μεταλλορίχη τελικά με τις διεκδικήσεις τους οδήγησαν σε μια συμφωνία που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ των ε, εργατικών ε, ενώσεων. Θα πρέπει να υπάρξει ανεξάρτητη έρευνα για τις για τις δολοφονίες αυτές. Και επίσης θα πρέπει να ικανοποιηθούν και τα αιτήματα των εργαζομένων για δίκες ε, συνθήκες εργασίας. Είναι τεράστια κοινωνική και οικονομική ανισότητα. Θα πρέπει να υπάρξουν απαραίτητα πρότυπα εδώ και προδιαγραφές και προστασία σε σχέση με τα εισαγόμενα προϊόντα. Τώρα, ε, ο κύριος Κατσμάρεκ η Νότιος Αφρική είναι μια χώρα με πολλές ιδιαιτερότητες. Είναι πλέον αναπτυγμένη χώρα και έχει θετική επιρροή προς τις γείτονες χώρες. Είναι φίλη χώρα προς εμάς και είναι απογοητευτικό να βλέπουμε ότι μια χώρα μπορεί να είναι τόσο επικίνδυνη Πολλοί είναι εκείνοι που φεύγουν από τη χώρα λόγω τη ανασφάλεια και πολλοί είναι που έχουν πέσει θύματα του καθεστώτο του Απαρτχάιντ παλιότερα. Τα θύματα του Αμερικανά θα πρέπει να πείσουν τι χώρε αυτέ να αναλάβουν ενεργό δράση όχι μόνο για να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά αίτια και να τιμωρήσουν του αυτούργου των δολοφονιών, αλλά για να περιοριστούν τα διορθωτικά σφάλματα μια τέτοια κατάσταση. Ε, το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσίων στα πλαίσια του οικονομικού απαρτχάιντ μας διευκολύνει να εντοπίσουμε τους ενόχους. Διαφθορά, εξαπάτηση, αυτή είναι η βασική λόγη και η χώρα αυτή είναι εκτεθειμένη στους κινδύνους του λαϊκισμού και της πολιτικής εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ Θέλω να εκφράσω την ε, συμφωνία με τον κύριο Τάνο και είναι πολύπλοκο το θέμα και φυσικά απερίφραστα καταδικάζουμε την σφαγή των 34 ανθρακορίχων, μια πολύπλοκη κατάσταση. Πριν γίνουν οι σκοτωμοί υπήρχαν δολοφονίες, επιθέσεις ε, στο προσωπικό ασφαλείας, στην αστυνομία και άλλους ανθρακορίχους. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν καταλήξουμε σε βιαστικά συμπεράσματα. Ο πρόεδρος Ζούμα και η κυβέρνησή του πιστεύω ότι έδρασαν όπως έπρεπε. Έκαναν αυτό που έπρεπε, πρέπει να περιμένουμε τώρα τι θα δείξει η δικαστική έρευνα, αλλά κυρίως να βρούμε τις ρίζες ε, της τραγωδίας και της όλης αναταραχής. Υπάρχουν κοινωνικο-οικονομικά αίτια τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επίσης, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριο Τάνοκ, θα πρέπει να βελτιώσουμε την δυνατότητα αστυνόμευση, συνεργασία με τους νοτιοαφρικανούς μας εταίρους. Δεν έχω ε, προσυπογράψει ε, γιατί ήμουν αντίθετος ε, στη λέξη σφαγή στον τίτλο γιατί μας οδηγεί σε βιαστικά συμπεράσματα και προτρέχει, προκαταλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνα που είναι σε εξέλιξη και είναι μια υποκειμενική πιστεύω ένα υποκειμενικό χαρακτηρισμό τη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριο Πάσκαν, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε. Τεράστια φτώχεια, τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Λίγοι πλούσιοι, πάρα πολύ φτωχοί. Και φυσικά αυτά προκαλούν κοινωνικές εντάσεις, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή στη Νοτιοαφρική. Τα γεγονότα του Αυγούστου στο ορυχείο Μαρικάνα ήταν ένα πολύ τραγικό γεγονός. Είχαμε βία καταστολή ε, της απεργίας από τους ε, αστυνομικούς με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Ήταν εκτεταμένα αυτά τα επεισόδια ε, και οδήγησαν και σε διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες και σε άλλες περιοχές. Το γεγονό ότι δεν κατέστη δυνατό να γίνει ένα ε, πολιτισμένος διάλογο με του ε, μεταλλορίχου για τι συνθήκε εργασία, αποτελεί και απόδειξη για το ότι οι πολυεθνικές φαίνεται να παραγνωρίζουν ε, το ανθρώπινο έργο και δεν εξασφαλίζουν αξιοπρεπεί συνθήκες εργασίας. Έχουμε ζητήσει να γίνει έρευνα, να, να υπάρξει απονομή δικαιοσύνης. Αυτό είναι το ελάχιστο. Το ελάχιστο μπορεί κανείς να διεκδικήσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της ο κύριος Μέρφη έχει το λόγο στα διεθνή μέσα ενημέρωσης έγινε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί σύγχυση για αυτό το θέμα, ε, ότι είναι ένα πολύπλοκο θέμα και ότι αφορά ε, τα συνδικάτα. Σε καμία περίπτωση όμως ε, δεν πρόκειται κάτι τέτοιο. Ήταν δίκαια απεργία των μεταλλορίχων για σωστό μισθό, για καλές συνδίκες εργασίας και ενώ έφευγαν κάποιοι τους περοβολούσαν στην πλάτη από την αστυνομία. Λένε πολλοί ότι ήταν προμελετημένη αυτή η σφαγή και κάποιοι θέλησαν να κατηγορηθούν ήδη με τα και ευτυχώ κατέπεσαν αυτές οι κατηγορίε. Ε, υπήρξε πραγματική προδοσία ε, των ε, αγώνων που έγιναν για την κατάργηση του Apartheid. και πρέπει να δούμε τις τεράστιες ε, ανισότητες και αδικίες που υπάρχουν. Μία μικρή ελίτ, ελάχιστη ελίτ η οποία ε, πλουτίζει σε βάρος ε, των πολλών που λιμοκτονούν. Θα είμαι παρόν και εγώ σε μία πορεία αλληλεγγύης που θα γίνει για την υποστήριξη μας προς τους διαδηλωτές και τους απεργούς. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τρεις ομιλητές. Καταρχήν η κυρία Φερχέμεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Οι διαμαρτυρίες από άτομα τα οποία οδήγησαν στα βία γεγονότα της 16ης ε, Αυγούστου και όπου υπήρξαν πολλοί τραυματίες είναι μια πολύ ε, ε, ε, ματηρή ε, περίσταση για τις την Νότια Αφρική που οφείλεται εις ε, την, ε, ε, τις κοινωνικές αδικίες και πρέπει να υπάρξει μία βελτίωση της αντιμετωπίσεως κρίσεων για τέτοιες έκτακτες καταστάσεις καθότι θα χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια για τις δυνάμεις ασφαλείας και έτσι έχει χαθεί και η νομιμοποίηση του ομολόγου του λαού και υπάρχει φόβος διαφθοράς γι' αυτό και θα πρέπει να εξετάσουμε και τις επιπτώσεις αλλά και τις αιτίες αυτών των γεγονότων. Χρειάζονται καλύτερες συνθήκες πλαίσιο κατά τις συζητήσεις των κοινωνικών εταίρων που πρέπει να είναι δίκαια και όλα αυτά ίσως έχουν λεχθεί ήδη αλλά πρέπει να στηρίξουμε τους ε, νοτιοαφρικανούς ομολόγους μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιακονσάρη έχει τώρα το λόγο τα πρόσφατα γεγονότα στην Νότιο Αφρική δεν πρέπει να θεωρηθούν σαν ένα μεμονωμένο γεγονός ε, απλώς ε, απικιοκρατίας αλλά αποτελούν ε, μία απογοήτευση και το αποτέλεσμα της δυσαρέσκειας. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η κυβέρνηση θα είναι στο ύψος των περιστάσεων και ε, θα εφαρμόσει τις ε, προτάσεις ε, και υποσχέσεις που έχει κάνει στο λαό και δεν θα υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ διότι υπάρχει αύξηση της φτώχειας, θέματα εργασιακά, και στην Νότια Αφρική πρέπει να υπάρξει μία μετατόπιση ε, του κέντρου βάρους προς ε, την ε, εφαρμογή μίας χρηστής πολιτικής όπως το είχε προβλέψει ο πρόεδρος της ΟΚΙΜΗ στην πρόσφατη πίσκεψή του στη χώρα αυτή. Ο κύριος Πρέτα. Ευχαριστώ. Με ανησυχεί ιδιαίτερω η κατάσταση στην Νότια Αφρική και είναι απογοτευτικό το πώ ε, κατέστηλε την διαμαρτυρία των Ανθρακορίχων η Προεδρία. Θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον ε, η... όλη αυτή η διαδικασία δεν αποτελεί μια παγίδα διότι κάποιοι ξεπερνούν το ρόλο του ως διαπραγματευτών για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αστάθειας και να αποκτήσουν πολιτική δύναμη. Είναι πολλοί παράνομοι εργαζόμενοι σε πολλά ανθρακοριχεία της Νότιας Αφρικής. Χθες, ε, μάλιστα, μπροστά στους ε, ανθρακορύχους ε, εκφωνήθηκε λόγος τον κύριο Μαλέμα που μας ανησυχεί με τις τοποθετήσεις του Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Πρώτος ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως υπόθηκε, πρόκειται για μια αποτροπιαστική τραγωδία. 34 ε, σκοτώθηκαν και κάποια αστυνομικοί δείχνει αυτό πόσο δύσκολο είναι να επιτύχει μια τεράστια μετάβαση από έναν ε, πολιτισμό και μια κουλτούρα βίας σε ειρηνικές ε, ε, καταστάσεις. Και ίσως θα πρέπει για αυτό το λόγο να δούμε και να συγκρίνουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Βέβαια, οι ανθρώπινες ζωές είναι ιερές, ιερές και κάθε θάνατος ε, είναι τραγικός, όποιος και αν είναι αυτός. Και όλα αυτά πρέπει να τα καταδικάσουμε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τρία πράγματα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν. Σε ένα υψηλότερο επίπεδο μπορούμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να φροντίσει να υπάρξει ομερή κατανομή του πλούτου της Νοτιοαφρικής. Δεύτερον, θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πίεση ιδιαίτερα στους επιχειρηματικούς κύκλους, ώστε οι εταιρείε οι ε, να αναλαμβάνουν και την κοινωνική ευθύνη που τους αναλογεί. Επίσης πιστεύω ότι η ηγεσία ε, των συνδικάτων σε διεθνές επίπεδο θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε τα ε, αντίπαλα εντό αγωγικών συνδικάτων να διεξάγουν τι δραστηριότητέ του ε, μέσα σε αστικέ δικαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κατσού για ένα λεπτό. Τα γεγονότα της Μαρικάνα είναι πραγματικά τα πλέον βία γεγονότα από τον τερματισμό του Απαρτχάιτ στην Νότια Αφρική. Θα πρέπει να δούμε με βλέμμα κριτικό την ε, εξέλιξη των κοινωνικών συνθήκων στη χώρα αυτή από το τέλος του Απαρτχάιτ και μετά. Θα πρέπει μετά το θάνατο των 34 ανθρακορίχων να σκεφτούμε το κατά πόσο να παρεμβαίνει σωστά η αστυνομία, η αστυνομική δύναμη στη χώρα αυτή, προκαλώντας τόσο βία γεγονότα. Επίσης, ε, ακόμη 50 περίπου ανθρακορίχοι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν έγινε καμία αντικειμενική έρευνα πριν τη δίκη. Θέλουμε λοιπόν να θυμίσουμε στο Αφρικανικό Συμβούλιο ότι εγγυήθηκε περισσότερη ευημερία για όλους τους Αφρικανούς ε, της Νότιας Αφρικής μετά το τέλος του Απαρτχάιντ. Αυτό πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε κυρία Γιάτερμάκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι ειδήσει που φτάνουν από την Νότια Αφρική, ο θάνατος των ανθρακορίχων είναι κάτι που μας συνταράσει. Πώς μπορεί κανείς να διανοείται ότι μια ειρηνική διαδήλωση, μια απεργία, τελικά καταλήγει σε ένα λουτρό αίματος που προκάλεσε η αστυνομία. Όταν είδα τις ε, εικόνες από τα ε, επεισόδια αυτά, Πραγματικά έφτασα να μην καταλαβαίνω τι βλέπω. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αληθινέ. Πίστευα ότι μπορεί να είναι πλαστέ, ε, παραπημένε. Τι κάνει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Νότια Αφρική για να υπάρξει ανεξάρτητη σοβαρή έρευνα. Η Λέδη Άστον θα έπρεπε να προσφέρει και την βοήθεια της Ευρώπης στην Νότια Αφρική με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες στο κοινωνικό κλίμα, να βελτιωθούν και να ηρεμήσουν οι κοινωνικές σχέσεις. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Είπατε εκπρόσωπος ε, και αντιπρόεδρος ε, και Αστόν επισκέφθηκε την Νότια Αφρική λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο αρχείο Μαρικάνα. Η τραγωδία δεν έπληξε μόνο την Νότια Αφρική. Σε ολόκληρο τον κόσμο πάρα πολλοί παρακολούθησαν αυτά τα δραματικά γεγονότα. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας για τις ζωές που χάθηκαν. Η κυρία Άστον συζήτησε την κατάσταση σε βάθος με τους νοτιοαφρικανούς αξιωματούς, του οποίου συνάντησε. Μεταξύ αυτών των προεξωτερικών των του Ζούμα. Προσφάτως εκλεγέντα Επίτροπο της Αφρικανικής Ένωσης. Χαιρετίζουμε τον ορισμό από τον πρόεδρο Ζούμα μιας ε, πλήρους ε, δικαστικής εξεταστικής επιτροπής η οποία θα διερευνήσει τα γεγονότα καθώς και τη σύσταση διεπιουργικής επιτροπής η οποία θα αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα μετά από την αιματοχυσία. Επίσης η κυρία Αστόν είπε στους ομολόγους μας από την Νότια Αφρική ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον και προσοχή και τις διαδικασίες και τα πορίσματα αυτής της έρευνας. Η Ευρωπαϊκή, μάλλον Επιτροπή που συγκρότησε ο πρόεδρος ε, Ζούμα θα έχει ως πρόεδρο έναν ε, πρώην πρόεδρο ε, του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας και αυτό είναι θετικό για τις προθέσεις του πρόεδρου Υπάρχει ε, στήριξη επίσης που παρέχεται στους πληγέντες, στις οικογένειες των θυμάτων και επιχειρείται να δοθεί μία λύση ε, στην ε, ρευστή και πολύ ασταθή κατάσταση που κρατήσει στον τομέα των ορυχείων. Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε και θα ήταν λάθος τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά είναι σημαντικό κατά την άποψή μας να δούμε ποια είναι τα βαθύτερα αίτια, αλλά να διευκρινιστούν και οι συνθήκες από τις οποίες έλαβαν χώρα τα γεγονότα αυτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχω... Έχω λάβει έξι ψηφίσματα. Θα κλείσει τώρα η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει μετά την ολοκλήρωση